στις 22 Τετάρτου 2010. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της 22 Τετάρτου 2010 έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν, άρα τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται. Έχω δύο ανακοινώσεις για το σώμα. Η πρώτη, θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι στη διάρκεια της παρούσας περίοδου συνόδου θα βρίσκονται στην Ολομέλη ορισμένοι επιπλέον τεχνικοί εικονοληψίας με ειδικό εξοπλισμό. Οι τεχνικοί αυτοί θα μαγνητοσκοπήσουν τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες μας με σκοπό την παραγωγή μιας ταινία πανοραμικής κάλυψης 360 μοιρών της διεξαγωγής των εργασιών του Κοινοβουλίου. Η ταινία αυτή θα προβάλλεται ως τμήμα της μόνιμης έκθεσης με θέμα της εργασίας του Κοινοβουλίου σε μια διαδραστική μακέτα της αίθουσας Ολομέλειας στο νέο κέντρο επισκεπτών στις Βρυξέλλες. Έχω λάβει σαφείς διαβεβαιώσεις ότι η παρουσία των τεχνικών θα είναι ιδιαίτερα διακριτική και δεν θα εμποδίσει κατ' ουδένα τρόπο τη διεξαγωγή των εργασιών μας. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Η δεύτερη ανακοίνωση. Έχω λάβει από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αιτήματα για τον ορισμό μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο κατάλογος των αλόγων ορισμών θα περιληφθεί στα συνοπτικά πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις μέχρι την έγκριση των συνοπτικών πρακτικών, οι ορισμοί αυτοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες προτείνω τις ακόλουθες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της Ολομέλειας αυτής της εβδομάδας. Την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, πρώτον η κοινή συζήτηση επί των δύο εκθέσεων του κυρίου Μέντες Δεβίγκο σχετικά με τη σύνθεση του Κοινοβουλίου θα αποτελέσει το πρώτο σημείο συζήτησης. Δεύτερον, στην ημερήσια διάταξη προστίθεται το νέο σημείο δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή σχετικά με την προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής τη 7 η Μαΐου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ, χωρί ψήφισμα. Το θέμα αυτό θα αποτελέσει το δεύτερο σημείο και προβλέπεται μόνο ένα γύρο ομιλητών από τι πολιτικέ ομάδε χωρί τη διαδικασία του Catch Τρίτον, ο τίτλος των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την τυποποίηση των ηλεκτρικών οχημάτων τροποποιείται σε δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά με οχήματα. Τέταρτον, η έκθεση του κυρίου Πρόντι, της οποία είχε προγραμματιστεί να γίνει σήμερα η συνοπτική παρουσίαση, μετατίθεται για απευθείας ψήφιση στην ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης. Αλλαγές για την πέμπτη τώρα. Πρώτον, η ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Μορέιρα σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία αναβάλλεται για την περίοδο συνόδου του Μαΐου 2. Δεύτερον, η ψηφοφορία επί της προτάσεως ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής περί καθορισμού κατευθυντηρίων γραμμών για τη συγκρότηση μηχανισμού αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς καθώς και περί κοινή προσέγγισης για την τιμολόγηση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποσύρεται από την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν παρατηρήσεις επ' αυτών αν όχι οι τροποποιήσεις εγκρίνονται και η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει και μία ε, πρόταση για αλλαγή στις ψηφοφορίες σήμερα. Ύστερα από τη χθεσινή συνεδρίαση μεταξύ του Προέδρου Μπούζεκ και του Προ... Πρωθυπουργού Θαπατέρο, συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να αρχίσει αμέσως ένας διάλογος στο υψηλότερο θεσμικά επίπεδο σχετικά με ορισμένες διαδικαστικές πτυχές που αφορούν την απαλλαγή του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, η Προεδρία προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του θέματος αυτού για προσεχή περίοδο συνόδου. Υπάρχουν παρατηρήσεις επ' αυτού. Θέλει καλής να σχολιάσει επ' αυτού. Δεν βλέπω χέρια. Θέλετε εσείς. Καθίστε κάτω. Εφόσον βλέπω ότι υπάρχουν παρατηρήσεις, θα ανοίξω τη διαδικασία για ένα ομιλητή υπέρ, ένα ομιλητή κατά. Ποιος θέλει να μιλήσει υπέρ της πρότασης. Υπέρ. Who wants to speak in favor of the proposal. Ο κύριος Σούλτς. Πρόεδρε, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ άκουσα για την ε, συνάντηση αυτή Μπούζα και Ζαπατέρο. Φαντάζομαι ότι πρόκειται για την ε, διευθέτηση των διαφιλονικούμενων ζητήματων ε, στην εκτέλεση του προπολογισμού του Συμβουλίου. Είναι τόσο λεπτής φύσεως που φαντάζομαι ότι είναι σκόπιμο να γίνει περαιτέρω συζήτηση. Οτιδήποτε θα αποφασίζαμε σήμερα εδώ θα ήταν ε, σκοπιμότερο να αποφασίσουμε να αναβάλουμε την ε, εξέταση της απαλλαγής. Εάν υπάρχει κάποια ευκαιρία, όπω είπαμε νωρίτερα, ζητήματα που έχουν μείνει ακρεμοί να λάβουν ικανοποιητικέ για το Κοινοβούλιο απαντήσει, θα πρέπει αυτή την ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε. Ταυτόχρονα αυτό αποτελεί και μια πρόσκληση προ το Συμβούλιο για ανοικοδόμηση εμπιστοσύνη, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση τη απαλλαγή, αλλά και για άλλου τομείς. Και έτσι υποστηρίζουμε την πρόταση. Ε, ένας ομιλητής ε, κατά, ο κύριος ε, voorzitter collega's ik heb de heer schulz goed aangehoord en ik ben. Eh, συνάδελφοι, άκουσα τον κύριο Σούλτ. Είμαι αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και ε, ήμουν και εγώ παρόν στι άτυπε συναντήσει με το Συμβούλιο. Η έκθεση που ζητείτε, τη οποία ζητείτε η αναβολή, έχει εγκριθεί με πλειοψηφία 27 ψήφων και 0 ψήφων κατά ή αποχής από την Επιτροπή ελέγχου του προπολογισμού. Είχαμε την δυνατότητα με τις άτυπες επαφές που είχαμε το Συμβούλιο να επιτύχουμε συμφωνία και συνένεση στην υπόθεση αυτή, αλλά το Συμβούλιο δεν συνεργάστηκε. Τώρα έρχεται το Συμβούλιο και μας δηλώνει τάχα πως είναι διατεθειμένο να διαθέσει κάθε ε, έγγραφο που απαιτούμε για την απαλλαγή. Επίσης πρέπει να σας πω ότι οι κανόνες μας ορίζουν ότι θα πρέπει τα έγγραφα να κατατίθενται σε κάθε περίπτωση εν ώψη της απαλλαγής στην άμεση του δημοσιονομικού κανονισμού, δηλαδή πριν από τις 15 Μαΐου του έτους νήσιν 1. Νήσιν 1 για την απαλλαγή του 2008 είναι όχι το 2010 αλλά το 2009. Μην ξεχνάμε επίση ότι έχουμε την προσεχή μας ολομέλεια τον, ε, Μα... τον ε, Μάιο, τέλη Μαΐου. Όχι αύριο λοιπόν, αλλά τέλη Μαΐου θα κληθούμε να ψηφίσουμε και νομίζω ότι αυτά όλα αποτελούν δείγμα πολύ κακής διαχείρισης των δημοσιονομικών μας. Ο μας, ο κύριος Τσαρνέτσκι, έχετε το λόγο. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Jestem szósty rok w Parlamencie Europejskim i είναι ο, έκτος μου χρόνος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα ήθελα παρόλα αυτά να φανώ διδακτικός ή να δώσω μαθήματα σε ιονδήποτε. Παρόλα αυτά θα ήθελα να μάθω από τον εισηγητή κάτι. Θα ήθελα να μας υπενθυμίσει ο εισηγητής ότι το κοινοβούλιο μας στα πλαίσια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, αυτής της κοινοβουλευτικής εντολής έχει ήδη δώσει το Νοέμβριο απαλλαγή στο Συμβούλιο. Το Νοέμβριο του 2009. Για μια ακόμη φορά λοιπόν το Συμβούλιο δεν παραδίδει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και εκπλήσωμε βαθύτατα από τη στάση του αυτή. Τώρα άρχισαν να μας δίδουν κάποια έγγραφα τα οποία αφορούν την περίοδο του 2007 είμαι έκπληκτος από τη συμπεριφορά του Συμβουλίου. Πέραν αυτού προσπαθώ να είμαι πραγματιστής. Προσπαθώ να βοηθήσω να καταλήξουμε σε κάποια συμβιβαστική λύση. Είναι λοιπόν τώρα η τελευταία ευκαιρία έτσι ώστε το Συμβούλιο να προετοιμάσει τα απαιτούμενα έγγραφα και να αποφασίσει να συμπεριφερθεί με υπεύθυνο τρόπο σαν όργανο. Ας δώσουμε λοιπόν δύο ή και έξι αν θέλετε το μέγιστο εβδομάδες προς το Συμβούλιο και να ψηφίσουμε τον μήνα Ιούνιο. Λοιπόν, της ψηφοφορίας όσοι είναι υπέρ ε, του αιτήματος της Προεδρίας για την αναβολή της ψηφοφορίας επί του θέματος αυτού για προσεχή περίοδο συνόδου, όσοι είναι υπέρ, τα χέρια σας παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και προχωράμε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρώτα, η έκθεση του κυρίου Γκαρσία Μαργάλο Ιμαρφίλ με ονομαστική κλίση ε, σχετικά ε, με την διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον ραπορτέρ. Ε, επόμενη έκθεση, έκθεση ΚΑΖΑ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου ε, προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στο ραπορτέρ. Η τρίτη έκθεση του κυρίου Σπερώνη σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Ράνστορφ. Την θέτω σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Σαρνέσκη σχετικά με την απαλλαγή ε, ε, του Γενικού Προπολογισμού τη ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα 4, δικαστήριο. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Τσαρνέσκη σχετικά με την απαλλαγή για το ελεγκτικό συνέδριο. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρίου Σαρνέσκη σχετικά με την απαλλαγή για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση κύριου κ. σχετικά με την απαλλαγή για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στο ραπορτέρ. Έκθεση τη κυρία Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση προπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτος 2008. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται έκθεση της κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2008 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του προπολογισμού της κοινωνικής υπηρεσίας ελέγχου της αλληλείας με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση τη κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση τη κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρία Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρία Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή τη Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Με ονομαστική κλίση. Σας επισημαίνω ότι υπάρχει ένα διορθωτικό το οποίο αφορά την ιταλική απόδοση της έκθεσης αυτής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση τη κυρία Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρία Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στην Θάλασσα. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρία Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Οργανισμού Εφοδιασμού της Euratom. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση τη κυρία Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωση και εργασία. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση τη κυρία Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή τη Eurojust. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού ως Frontex. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρία Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή της κοινή επιχείρηση για το ΙΤΕΡ και την ανάπτυξη της πυρηνική σύνδεξη με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρία Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή της κοινή επιχείρηση ΣΥΖΑΡ με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στη ραπορτέρ. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφορία της έκθεσης του κυρίου Σίμψον σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υποπίεση. Εξετάζουμε την πρόταση οδηγία. Τροπολογία 66. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, άρα καταπίπτει το μπλοκ νούμερο 2 Ποιοι είναι υπέρ της ε, πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι, ποιοι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και με ονομαστική κλίση I said that block two lap, lap in translation. Σα είπα ότι πρόκειται περί μεταφραστικού λάθου, οπότε παρακαλώ να κάνετε μαθήματα ξενογλωσσών θα τα, θα τα χρειαστείτε, θα τα χρειαστείτε για να μάθετε ελληνικά και να παρακολουθείτε τι στη χώρα επομένω. Ψηφίσαμε από τι ε, τροποποιηθήσεις πρόταση, ποιοι είναι υπέρ αυτή τη τροποποιηθήσεις πρόταση, τέλεια, κατά, αποχέ, γίνεται Και τώρα η νομοθετική πρόταση με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει από τη εκθέσεω του κυρίου Λάικτφριντ σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια τη πολιτική αεροπορία. Ψηφίζουμε μία σειρά τροπολογιών από την Επιτροπή. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 29. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τσεκ τροπολογία 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας Εγκρίνεται. Τροπολογία 44 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 45 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ε, η ψήφος ε, για την πρόταση όπως τροποποιήθηκε, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με ονομαστική ψήφο το σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στο ραπορτέρ. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία τη έκθεση του κ. Σίμψον σχετικά με του κοινοτικού προσανατολισμού για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Τροπολογίε 1 και 2 από την Επιτροπή. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνονται. Με ονομαστική κλίση η τροπολογία 3. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, η, πρόταση επί της, ε, η ψήφος της ε, πρότασης όπως έχει τροποποιηθεί ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με ονομαστική ψήφο η ψήφος επί του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στο ραπορτέρ. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Κυρίλοφ σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση. Μία σειρά τροπολογιών από την Επιτροπή. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 19. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψήφος επί της πρότασης ως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ψήφος επί του ψηφίσματος του νομοθετικού με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον ραπορτέρ. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τις συνέπειες της έναρξης ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα στι τρέχουσε διοργανικέ διαδικασίε λήψη αποφάσεω Omnibus. Σα επισημαίνω ότι η τροπολογία αριθμό 1 έχει αποσυρθεί. Άρα ψηφίζουμε επί του. Ε, με συγχωρείτε, ο κύριος έχει το λόγο. δευτερόλεπτα επεξήγηση απόσυρση της τροπολογίας μας. Αποσύρωμε λοιπόν την τροπολογία μας έχοντας απόλυτη και βάσιμη πεποίθηση ότι η διάσκεψη των Προέδρων, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα, θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της το πνεύμα και το περιεχόμενο της τροπολογίας μας. Υπενθυμίζω ότι η τροπολογία μας ζητά, όπως η Κομισιόν, μελετήσει την αλλαγή του κανονισμού για το απευθείας εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις περιοχές της Κύπρου που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ε, ψηφίζουμε ε, τώρα την παράγραφο 1, ε, σημεία 4 έως 9 ε, του αρχικού κειμένου. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές. Ε, θα το ελέγξω ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψήφος επί της, ε, του ψηφίσματος συνολικά. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Σάιερ σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Α, καταπίπτει, με συγχωρείτε. Η τροπολογία 6 καταπίπτει. Πηγαίνουμε τώρα και καταπίπτει και το αρχικό κείμενο. Πηγαίνουμε τώρα στην τροπολογία 3. Τροπολογία 3 λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, η τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. As I noticed that the socialist group seems to be η σοσιαλιστική ομάδα αργεί να σηκώσει τα χέρια της. means abstention. Okay? So when you hear Λοιπόν, όταν ακούτε υπέρ στα ελληνικά, σηκώστε τα χέρια σας έτσι κι αλλιώς. <laughs> Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία τις έκθεσεις του κυρίου Βαντάλεν σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απογύπτεται; Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το αρχικό κείμενο παραγράφου 8 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η σοφορία. Πέρες σοφορίας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο παραγράφου 30. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος επί του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης κυρίας Τρούπελ σχετικά με την Γιουροπεάνα, τα επόμενα βήματα. υπάρχει μία τροπολογία, τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο επομένως καταπίπτει. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης της κυρίας Πόλσεν σχετικά με την αξιολόγηση και αποτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 9 σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο μέρος με ονομαστική κλίση. Roll call vote on the third part. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 18 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 19 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Recital C. Σε δύο μέρη. Check what. Recital C. Τη λογική σκέψη γάμα. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος επί του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Η ρίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Λεφόλ σχετικά με τη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κλιματική αλλαγή. Η παράγραφος 7 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 8 σε δύο μέρη, ε, με συγχωρείτε, η παράγραφος 18 σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία στο δεύτερο μέρος. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 20 σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 31 σε τρία μέρη και τα τρία με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ο, μισό λεπτό. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 36 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Citation 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα σοφορίας, Εγκρίνεται. Τελική ψήφος επί του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Λεφόλ. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία από τις έκθεσεις του κυρίου Ντόρφμαν σχετικά με την γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Η παράγραφος 5 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος στο δεύτερο μέρος παραγράφου 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τελική ψήφος. You want to check on 6. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην παράγραφο 6. Άρκετη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Ντόρφμαν. Η μερίσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία τη έκθεση τη κυρία Τελκαστή Βέρα σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. Η παράγραφος 14 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελ... Check. I'll take three checks today. If I'm right in all three, I take no more. Αν έχω δίκιο σε αυτό, δεν θα ακούσω άλλη. Ηλεκτρονικά. Άρκετη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Είχατε απόλυτο δίκιο. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Τερκαστήλιο Βέρα. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Λιμπεράτσκι σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του Γενικού Προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα 3. Ε, Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί. Ο κύριος Λιμπεράτσκι, ο εισηγητής, έχει το λόγο. Δεν είμαι ο κύριος Λιμπεράτσκι, αλλά αν μου επιτρέπετε θα κάνω μια τεχνική διόρθωση στην 248 παράγραφο. Πρόκειται για, τους, για τις μονάδες 1 έως 4 του εργοστασίου του Κοσλοντουή. 1 έως 4. Θα εξεταστούν όλες αυτές οι παρατηρήσεις για την ακρίβειά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι θέλει ή δεν θέλει το λόγο. Ναι, τον έχετε. ευχαριστώ για τους συναδέλφους που πήραν μέρος στη συζήτηση αυτή. Η διαδικασία απαλλαγής δεν αφορά τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και τα ίδια τα κράτη-μέλη φυσικά, τα οποία αντιπροσωπεύει το Συμβούλιο. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξουν κάποιες προτάσεις οι οποίες να μας οδηγήσουν στο μηδενικό λάθος. Να υπογραμμίσουμε τα προβλήματα τα οποία βρίσκονται πάντα σε εκκρεμότητα και να συνδυάσουν τις προσπάθειες που κάνει και το ελεγκτικό συνέδριο και εμείς έτσι ώστε να εντοπίζουμε στο μέλλον άμεσα τους προβληματικούς τομείς. Με τη νέα συνθήκη, τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η ίδια η διαδικασία απαλλαγής. Η έκθεσή μου λοιπόν ζητά να υπάρξει μια συζήτηση υψηλού επίπεδου ανάμεσα στα όργανα και ανάμεσα στις χώρες μέλη που είναι ουσιαστικά υπεύθυνοι για τη διαχείριση του 80% των δαπανών. Αναφέρομαι ε, στην απαλλαγή του 2008. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία ισχύουν και για σήμερα και η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα του παρελθόντος και θα πρέπει τα, οι πιστώσεις οι οποίες θα είναι διαθέσιμες να χρησιμοποιηθούν με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεν θα πρέπει να αλλοιωθεί η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες όπως, όπως η Τουρκία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έξυπνα τα χρήματα αυτά και να ωφεληθούν οι πληθυσμοί των χωρών μας και μέσω της χρήσης των διαφθορτικών ταμείων. Προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο τις επόμενες εβδομάδες έτσι ώστε να κακοφορήσουν οι προτάσεις τις οποίες κάνω και ελπίζω να επανέλθω στα πλαίσια της εφαρμογής των αποφάσεων αυτών τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ, κύριε Λιμπεράσκη. Προχωράμε τώρα στην ψήφο. Το σύνολο της πρώτας απόφασης με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Προχωράμε στην δεύτερη απόφαση αναφορικά με την εκπαίδευση κλπ. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτη απόφαση Τελεστικός Οργανισμός για Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα. Είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέταρτη απόφαση. Executive Agency for Health and Consumers. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέμπτη απόφαση. Trans-European Transport Network Executive Agency. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Προχωράμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 17. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Ποιοι είναι υπέρ. Not here. 18. Is it in two parts? Με συγχωρείτε. Η τροπολογία 18 είναι σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος τροπολογίας 18. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος τροπολογίας 18. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Δεν σηκώνει κανείς τα χέρια του. Τροπολογία 12. Amendment 12. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία με συγχωρείτε, αρχικό κείμενο. Δεν καταπιπτεί, είναι διαφορετικά. 54 οι υπόλοιποι σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Με ονομαστική κλίση. Με συγχωρείτε. Με ονομαστική κρίση τροπολογία 2. Άρκετη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η παράγραφος 116 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 9 και 14 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας φοβορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 σε δύο μέρη συμπεριλαμβανομένου και του όρα λαμμένου που υπάρχει. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 10 και 15 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Η τελική ψήφος επί του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. It's roll call. νέο ναι, ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Λιμπεράτσικη. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία τη έκθεση τη κυρία Αγιάλα Σέντερ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού του 7ου, 8ου, 9ου και 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη για το οικονομικό έτος 2008. Ε, η ψήφος επί της απόφασης ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα η τροπολογία στο νομοθετικό ψήφισμα. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και η, τροπολογία 2 καταπίπτει. Επομένω, η τελική ψήφος επί του νομοθετικού ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στη ραπορτέρα. Η μερίστη διάθεση προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Στάες σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση γενικού προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τμήμα 1. Τροπολογίες 4 και 37. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Is, is that Με συγχωρείτε. Δικό μου λάθος, δικό μου λάθος. Η ψήφος, η ψήφος επί της αποφάσεως συνολικά με roll call vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στι τροπολογίε επί του ψηφίσματο, τροπολογίε 4 και 37. Ποιοι είναι υπέρ είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση. Παρακαλώ έχετε το λόγο για την, ε, για την ε, προφορική τροπολογία. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Θα θέλαμε να καταθέσουμε μια προφορική τροπολογία στο πρώτο τμήμα της συγκεκριμένης τροπολογίας. Θεωρούμε ότι μια σωστή διακυβέρνηση, στα πλαίσια μιας τέτοιας διακυβέρνησης, το management παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να επιλέγονται με σωστό και αξιοκρατικό τρόπο. Και να προσθέσουμε επίσης εδώ, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ισορροπία και τις ίσες ευκαιρίες ανδρών γυναικών. Στην ουσία εισάγουμε δύο στοιχεία, ίσες ευκαιρίες από τη μία, γεωγραφική ισορροπία από την άλλη. Ονομαστική κλίση επομένως στο πρώτο μέρος της τροπολογίας 6 συμπεριλαμβανομένης και της ε, προφορικής τροπολογίας. Α, με συγχωρείτε. Εάν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία, από 40 βουλευτές μπορείτε να σηκωθείτε. Δεν είναι αρκετοί βουλευτές, άρα ισχύει η τροπολογία και προχωρώ τώρα στην ψήφιση. Δεν είναι ανοιχτό για πάντα, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ. We are voting on the Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 6 με ονομαστική κλίση. Συμπεριλαμβανομένης της προφορικής τροπολογίας υπέρ παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Για διευκρίνηση, ψηφίσαμε την έκτη τροπολογία με ή χωρίς την προφορική, παρακαλώ. Πάντα ήμουν σαφής, σαφής με το oral amendment. Το πρώτο μέρος της 6 εγκρίθηκε με το oral amendment. Δεύτερο, Αγαπητοί συνάδελφοι, ζητήθηκαν 40 άτομα τα οποία έπρεπε να σταθούν και αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε περιόριστο χρόνο για να σταθείτε. Έγινε το αίτημα, δεν σηκώθηκαν 40, κάποιοι σηκωνόντουσαν, καθόντουσαν. Λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε, αλλά πρέπει ο Πρόεδρος να κάνει να λάβει μια απόφαση. Πλην όμω, εάν θεωρείτε ότι επικράτησε κάποια σύγχυση και αν δεν υπάρχει πρόβλημα με τον κανονισμό, να το ξαναπώ. Πρώτο τμήμα συμπεριλαμβανομένη τη προφορική τροπολογία ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα συμπεριλαμβανομένη τη προφορική τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. The vote is closed. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος, ε, ε τροπολογία 10. Αμε συγχωρείτε. What happens now, does it fall? Does, then 10 and 42 fall. I'm τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 9 και 38. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 31 σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Οι τροπολογίες 10 και 42 καταπίπτουν. Τροπολογία 32 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 13 και 39. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 15. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Τροπολογία I will do it because I made a mistake before, but I think that was my last mistake. Φαντάζομαι ήταν το τελευταίο σφάλμα αυτό. 6. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 σε δύο μέρη και τα δύο με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το αρχικό κείμενο της παραγράφου 86 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 34 και 41 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Πάλι. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τριάντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τελική ψήφος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια. Η επόμενη έκθεση του κυρίου Τσαρνέσκη, όπως αποφασίστηκε σήμερα, αναβάλλεται. Και περνάμε στην έκθεση του κυρίου Τσαρνέσκη σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά το τμήμα 6, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η ψήφος επί του της συνολικής απόφασης. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στο ψήφισμα τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος επί του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Τσαρνέσκη, τμήμα 7, Επιτροπή των Περιφερειών. Ψηφοφορία επί του συνόλου της αποφάσεως. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στο ψήφισμα τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψήφος επί του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκθεση Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή, απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχο των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ονομαστική ψήφο η ψήφος επί του ψηφίσματος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια. Έκθεση της κυρίας Μάθιου για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Με ονομαστική κλίση η ψήφος επί της απόφασης άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με ονομαστική ψήφο η ψήφος επί του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια. Η μερίσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία τη έκθεση του κ. Σαλαφράνκα σχετικά με τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι σχέσεις με τη Λατινική Αμερική. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η κυρία Γιάλα. Ε, Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν ψηφίσαμε την απαλλαγή για την κοινωνική και οικονομική επιτροπή. Ίσως κάνω λάθος. Περάσαμε απευθείας στην Επιτροπή των Περιφερειών. Τι δεν κατάλαβα καλά. Επαναλαμβάνω, τροπολογία 20. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Let me repeat my kind request to the... Να επαναλάβω το αίτημα μου παρακαλώ προς το σοσιαλιστική ομάδα να σηκώνουν τα χέρια τους. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Ναι, τροπολογία 11 εννοώ, με συγχωρείτε. Τροπολογία 11 στην παράγραφο 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο καταπίπτει. Τροπολογία 24. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται 14 Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 24 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. This is my second victory, I believe, in a row. Δεύτερη μου νίκα, νίκη στη σειρά από ό,τι φαντάζομαι. Παράγραφος, τροπολογία, με συγχωρείτε, 16. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 29 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 48. Αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Χιν Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 32. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επομένως καταπίπτει το, αρχικό κείμενο της 55. Παράγραφος 56, αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 58. Αρχικό κείμενο. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψήφος επί του ψηφίσματος ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Σαλαφράγκα Καταλάβατε ότι κάνουμε τις ψηφοφορίες μιας ολόκληρης εβδομάδας του Στρασβούργου σε ένα απόγευμα στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ για την επομονή και την επιμονή που δείχνετε. Προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την προσεχή διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά της 5ης Μαΐου 2010. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Α, νομίζω απορρίπτεται αλλά το ελέγχω. Ηλεκτρονική ψήφος για την τροπολογία 7. Πέρας σοφορίας. Απορρίπτεται το αρχικό κείμενο της παραγράφου 2 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Με ονομαστική κλίση. Άρκετη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται.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 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέμπτο, πέμπτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Πρώτο μέρος της τροπολογίας 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Check the first part of amendment 2. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 2 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έξι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ψήφωση τελική επί του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι άλλες προτάσεις καταπίπτουν. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία των δύο προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με το SWIFT. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ο κύριος Άλμπρεκτ ζητάει το λόγο για ε, τροπολογία 8. Κύριε Άλμπρεκτ, έχετε το λόγο. Uh, ναι, θα παρακαλούσα, ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η τροπολογία στην παράγραφο 8 της Γκουε και των Πρασίνων είναι ίδια διατύπωση με το ψήφισμα του Σεπτεμβρίου 2009. Είναι ακριβώς η ίδια. Θα ήθελα να σας ενημερώσω μόνο γι' αυτό. Είναι ακριβώς η ίδια θέση και δεν πιστεύω ότι υπάρχει αλλά, ε, να αλλάξει οτιδήποτε πριν τις διαπραγματεύσει για το SWIFT. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Άλμπρεκτ. Ψήφο Επιστροπολογίας 8 Η ραπορτέρ ζητάει το λόγο. Κυρία Πλάσορτ. Θα ήθελα να πω στους αδέλφους ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου η θέση μας. Το ψήφισμα ε, είναι δεδομένο και η τροπολογία αυτή περιττή. Ευχαριστώ. Τροπολογία 8. No, we cannot have a debate on this issue. Δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα. Well, I'm sorry. Uh, Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Αισθάνομαι έτσι μεγάλη γενναιοδόρια σήμερα. Δέκα δεύτερα, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω μόνο ότι είναι σημαντικό. Και να μην με ενοχλούν οι συνάδελφοι της ακροδεξιάς, παρακαλώ. Και εσείς θέλετε να είστε ενήμεροι, πιστεύω, για το θέμα, έτσι δεν είναι. Περί τίνος πρόκειται. Ε, σοριδών ε, αποστολή ε, προσωπικών δεδομένων στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ναι ή όχι. Αυτό είναι η τροπολογία 8. Υπέρ ή κατά, τουλάχιστον να ξέρετε περί τίνο πρόκειται. 8. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ψήφος επί του τελικού ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουν απομείνει δύο μόνο ψηφοφορίε. Κουράγιο, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ψηφοφορία τη πρόταση ψηφίσματο έξι πολιτικών ομάδων σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίε σχετικά με τι καταστάσει ονομάτων επιβατών PNR. Τροπολογία 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δέκα, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εννέα, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έντεκα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δέκα έξι, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Τέλος. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία των τεσσάρων προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόριξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της οφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η τελική ψήφος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε 21 αιτήσει για επεξήγηση ψήφου. Την πέμπτη αυτά. Ευχαριστώ πολύ.